παρατηρήσει σε σχέση με τα πρακτικά θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά. Στι 9 Δεκεμβρίου 2008 ο κύριος Βίτολ Τσόμτσακ έχει κάνει μια αίτηση για την διατήρηση της κοινοβουλευτικής του ασυλίας και των δικαιωμάτων του σε σχέση με μια νομική διαδικασία που λαμβάνει η χώρα στην περιοχή Οστροφ Κοπόσκι. Το Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφράσει την άποψή τη για το θέμα αυτό τον Απρίλιο του 2006 και επίση τον Φεβρουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2008. Θα ζητηθεί η γνώμη τη Νομική επιτροπής. Ο πρόεδρο τη Νομική επιτροπής έχει ζητήσει εξ ονομάτων τη Επιτροπή του οι τέσσερι αιτήσει ε, άρση ασυλία του κ. Χέρν Τόμτσακ να θεωρηθούν απαράδεκτε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων στις 11 και 12 Φεβρουαρίου